χαίρετε. Πρώτα απ' όλα να σας κάνω μια ανακοίνωση. Μετά από διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες θέλω να ενημερώσω το σώμα για τις εξής προτάσεις για αλλαγή στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης. Η συζήτηση για την προφερική ερώτηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων συμφωνίας ελευθερών εμπορίου με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θα καταλήξει με ένα ψήφισμα που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου την πρώτη ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Υπάρχουν αντιρρήσει. Ο κύριο Σόλτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαστε κατά της ψηφοφορίας και σε συμφωνία με τους βασικούς εισηγητές, τον κύριο Μπερντλάνι και τον κύριο Κασπάρη, προτείνουμε να ψηφίσουμε στη δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι ε, χρήσιμο να υπάρξει τέτοια ε, επιταχυμένη διαδικασία. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρο, ωραία να ψηφίσουμε την πρόταση για το Φεβρουάριο 2. Ποιοι είναι υπέρ του να γίνει η ψηφοφορία στη δεύτερη σύνοδο του Φεβρουαρίου. Κατά, αποχέ, ωραία, εγκρίνεται. Να περάσουμε τώρα στι ψηφοφορίες. Δεν έχουμε πολλέ. Έκθεση του κυρίου Μωράιες για την αυτοπομεμένη ανταλλαγή στοιχείων για τις άδειες κυκλοφορίες οχημάτων στη Λετωνία. Ονομαστική ψηφοφορία η οποία και άρχεται.